Dear colleagues της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, να συνεχίσουμε. Μας απομένουν πολλές ακόμα ψηφοφορίες. Δεν θα ψηφίσουμε για το 11. Θα ξεκινήσουμε με το 16. Γιατί ο αντιπρόεδρος κ. Λούνατσεκ μου ζήτησε χτες να ξεκινήσουμε με αυτό. Διότι έχει να πάρει ένα αεροπλάνο για την Αυστρία. Ε, Ούλρικε, έχεις να πεις κάτι. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε αυτή τη μικρή αλλαγή στην μέση διάταξη. Ως ηγήτρια για το κοσυφοπέδιο, ε, χαίρομαι που έχουμε αυτή την ψηφοφορία για τις Γενικές Αρχές για τη Συμμετοχή του κοσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου. Πολύ σημαντικό βήμα για να έρθει το Κωσυφοπεδίο πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πολιτιστικά θέματα, για τα οποία μόλις ψηφίσαμε. Ε, ε, τεχνικά θέματα, επιστημονική συνεργασία, περιβαλλοντική συνεργασία και δεσμούς κλπ. Επίσης, για ορισμένα αυτά τα προγράμματα θα συνεισφέρει το κοσυφοπαίδιο στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ, είναι σημαντικό βήμα στη διαδικασία ε, ολοκλήρωση και ένταξη του κοσυφοπαιδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και χαίρομαι που ε, έχουμε σημαντική υποστήριξη σε αυτή, την αυτή τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, λέει ο Πρόεδρο, περνάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται. Λίγη. 45 υπέρ, 8 κατά. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο θέμα, ε, διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Ο κ. Φανόρτεν, εισηγητής. Τζέφρι, θες να πεις κάτι? Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιοδησηγητές ε, για τη συνεργασία τους. Ε, ελπίζω ότι θα ακολουθηθούν οι, οι οδηγίες που έχω δώσει για την, τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ξεκινάμε. Συμβασμός υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση παριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 12 και Ντονζόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 32 κατά 29 υπέρ. Συμβαστική πρόταση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 34 υπέρ κατά καποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την, το σχέδιο γνωμοδότησης άρχεται δύο ακόμα που δεν έχουν ψηφίσει ένας λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 54 υπέρ 6 κατά Συγχαρητήρια κύριε Σίγητα. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Σημείο παριθμών 12. Συγκρότηση ενωσιακού συστήματο ελέγχου των εξαγωγών τη μεταφορά τη μεσητεία, τη τεχνική βοήθεια και τη διαμετακόμιση ειδών διπλή χρήση. Ε, Μαρέτσιε Σάκε, η θε να πει δύο λόγια. Όχι. Δυστυχώς δεν έχω μπροστά τον κατάλογο. Ορίστε τον βρήκα. Τροπολογία. Όχι, 39 είναι μη παραδεκτή. Ξεκινάμε μια εξαιρετική ε, τροπολογία. 40, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ σοφή η απόφασή σας. 41. Άλλη μια εξαίρετη. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Γιατί είπε δύο. Με εκπλήσω. Περνάω στη συμβαστική παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμόν 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται να το ελέγξουμε τη 47 άρχεται η ψηφοφορία λίγη Πώς μου το κάνετε αυτό 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη συμπεριφορά σας. Απορρίπτεται προφανώς. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω διαφορά, αλλά σε παληθεύσουμε. 60. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 45 κατά 18 υπέρ. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Επαλήθευση για την 61. Άρχεται. Λίγη. 32 υπέρ 28 κατά. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 και 69 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Όχι, 13 υιοθετήθηκε, άρα καταπίπτει η 70. 71 και 72 υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και οι δύο. 14 υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 και 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση 93. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 της κυρίας Λόζινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 104 Λήξη ψηφοφορία 40 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται Τι δεν δουλεύει? Το μηχάνημά σας. Ωραία, έρχεται αμέσως ο τεχνικός. δεν έτσι κι αλλιώς δεν θα κάνει καμία διαφορά, έτσι δεν είναι. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε την 106. Λήξη τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω τι ψηφίζει το ΕΛΚ. Ας επαληθεύσουμε την 118 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτεται και αυτή. 120 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και πάλι επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε. Την 21. Έναρξη. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 138 137 υπέρ κατά εποχέ. απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 επαληθεύουμε έναρξη της ψηφοφορίας Λήξη. Σαφώς απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 139. Λήξη. Πολύ μικρή διαφορά, αλλά απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Άλλη μία από τον David Μάρτιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 λήξη εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με τις τροποποίησεις άρχεται. λίγη. Εγκρίνεται 49 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Στην εισηγήτρια μάλλον. Περνάμε στο σημείο 13. Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας περιλαμβανομένης της γενοκτονίας. Εισηγητής ο κύριος Πρέντα. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Πρέντα. Ας περάσουμε στις υποφορίες. We start with... Ξεκινάμε με τη συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολύ μεγάλη, πολύ και λύσο κατάλογος, δυστυχώς. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να κάνουμε έλεγχο. εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, παρέθηκα, ας κοιτάξουμε. 76, ας ελέγξουμε, ε, η άρχεται ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά,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 Περιέργως εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού είναι η 80. Α, να τι; Ναι, κατά τμήματα ψηφοφορία. 80 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82ο τμήμα έλεγχος για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπει ένας συνάδελφος. εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 120 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 προς 26 εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 επερ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 επερ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 επερ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 επερ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 επερ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 153. 154 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. 155, 167 και 171 υπέρ κατά εποχε απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 156 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 23 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 176 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 Α, εγκρίνονται αυτά, καταπίπτουν, άρα συμβαστή 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. 27. Τροπολογία 27 του κυρίου Κοράου. Όχι καταπίπτει. Την κρίθηκε 13. Όχι. Ναι. 28. 28 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά, εγκρίνεται. Στην τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από την 47 μέχρι πού θέλετε μπλοκ. Από την 47 ως την 54 ψηφίζουμε μπλοκ. Υπέρ, κατά, αποχές. Όλες εγκρίθηκαν. Ένα, υπέρ. Μπλο... Να, αφήστε με να ελέγξω πρώτα πριν το μπλοκ. Ένα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα υπάρχει αίτημα για να ψηφίσουμε ε, συνολικά από κοινού από την 4 στη 12. Η κυρία Λοχμπίλερ αρνείται. Η κυρία Λόιζινγκ λέει όχι. Δεν θέλω άλλες ε, διαταγές από τη γερμανική πλευρά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 Πέρα, Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το ψήφισμα που τροποποιήθηκε. Έρχεται η ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι μας λείπουν. Ένας. Ψηφίστε. Κλείση ξυπνήματος για την Ευρώπη. 50 προς 2 συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα, στον εισηγητή. Σημείο 14. Σύσταση προς το Συμβούλιο για την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εισηγητή, ο εγκεκριμένο συνάδελφο κ. Κόβατσε. Θέλετε να πείτε κάτι. Τι κρίμα. Να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 του κυρίου Πάετ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Δύο μας λείπουν πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 54, κυρία Λοχμπίλερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Κόβατσεφ Πρέντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίθηκε. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. απόχέ Να ελέγξουμε την 75. Απορρίφθηκε. 74 υπέρ. Κατά αποχές. Καμία αντίδραση από αρκετέ ομάδες. Να ελέγξουμε και πάλι. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 76 υπέρ. Κατά. Αποθέσει εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές 83 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Ένας τεχνικός. Κύριε, Εν τω μεταξύ το φτιάξει ο τεχνικό. 83 υπέρ. Τα χεράκια. Κατά. Πώ ψήφισαν οι φιλελεύθεροι. Υπέρ. Οπότε λέμε ότι εγκρίνεται. Τώρα δουλεύει το μηχάνημα. Τι κάνατε. Α, η αριστερή πλευρά της οθόνης λειτουργεί όχι δεξιά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, μετρήσαμε σωστά. Για προς στιγμή προσμετρώνται οι ψήφοι. 83. Ναι, αλλά τώρα δουλεύει πάλι το μηχάνημα. 83. Λείπουν τρεις συνάδελφοι. Ωραία, Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με 30 προς 28. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 έλεγχος. Ωραία. Να ελέγξουμε ξανά. 85. Πέρας. 28 προς 28. Μεσοψηφία. Απορρίπτεται. Πολύ κοντινά αποτελέσματα στη διαφορά. 86 πέρα. κατά εποχές Απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο. Εντάξει. 90 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Με σαφή διαφορά. Κάνα πρόβλημα. Το μηχάνημα καμιά φορά δουλεύει κιόλα. 89. Τάνο και πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Λόχμπιλερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές 93 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 101-114 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνονται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 116-117 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 118-119 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132-133 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136-137 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 141 έλεγχος. 140 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 100 κατά πίπτη. 144 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 145-146 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Εντάξει λοιπόν. 145-146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκαν του κυρίου Καστάλλου τώρα υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, ωραία λοιπόν, 142. Τρεις λοιπόν, ωραία πέρας. Εγκρίθηκε. Τα βλέπετε καλά από εκεί. 147-148 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Έλεγχο. Το φοβόμουν θα συμβεί. 147-148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 11. Επέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 155. Τάνοκ. Επέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156. επέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157. Εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι απορρίφθηκε. Έλεγχος. Όχι. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίβεται. 180 υπέρ, κατά, έλεγχος. 180. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 προς 24. Αργήσατε, αλλά δεν πειράζει, πάλι τα καταφέρατε. Που είμαστε 178 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνονται. 185, 170, 195. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απολύτω. 13 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 193 μίλαν μόνο. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Εποχέ. απολύτω. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 θέλετε έλεγχο. Ωραία λοιπόν, ζητήθηκε να ελεγχθεί από τους πρασίνους. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Δύο δεκαεννέα Μποργέτσιο υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 221 και 222 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. 227. Να ψηφίσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Δύο ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι φιλελεύθεροι πρέπει να ε, μα δείχνουν σαφέστερα τι ψηφίζουν γιατί αυτοί αποφασίζουν τελικά. 2-32 υπέρ. Και τι κάνουν τώρα οι φιλελεύθεροι. Α, είναι υπέρ. Ωραία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Κοιτάζω μόνο του φιλελευθερου τώρα. τώρα. 2-30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ελέγχουμε τη 2.31 Πέρας, εγκρίνεται. 2.33 line υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γκόμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.54 και 55 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα των 2.54 και 55. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.47 Λάινεν Post Μπροκ Κόβατσοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3, 7 και 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 4, 10, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 8 άρχεται πέρας Εγκρίνεται. 14 καταπίπτει, 9 λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το 18 του κυρίου Λάινεν. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 λόχπιλερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27-28 υπέρ κατά αποχές. Σοσιαλιστές είναι κατά, τότε απορρίπτονται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 του κυρίου Πρέντα. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε άρχεται. Πέρας. 45 ε, ε, υπέρ 4 και 9 αποχές εγκρίνεται. Δυστυχώς φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία. Το 15. Το πλαίσιο επανεκατάσταση της Ένωσης. Μετεκατάσταση, κατάσταση της Ένωσης. Θέλετε να πείτε τίποτα. Αρχίζουμε με τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε στην τελική ψηφοφορία. Πάμε στο 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Το 74. Νομίζω πως ήταν σαφές ότι ήταν υπέρ το αποτέλεσμα, αλλά ας ελέγξουμε. Στην 74 είμαστε. Ελέγχουμε την 74 παρακαλώ. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Και ένας. Ένας δεν τα έχει καταφέρει. Εγκρίνεται 30 με 24. Εγκρίνεται λοιπόν 74, οπότε 76, Σαφχάουζε και άλλοι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ο... Άλλη μία, 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 παντζέρι υπέρ κατά αποχές η είναι υπέρ τότε κρίνεται 82 βαλέρο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85-86 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Πέρας εγκρίθηκε. 91-92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται επίση. 96 και 7 και 98 ε, υπέρ, κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εγκρίνεται μάλιστα. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Αν να ελέγξουμε την 102 είπατε. Καλά, ελέγχουμε την 102 της κυρίας Βεργιά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 23 ε, υπέρ 31 ψηφί κατά. Απορρίπτεται. Σαφώς ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 105. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Μα μόλις ε, κέρδισε την τροπολογία της αυτή η κυρία Βεωζιά. 106. Πώς. Α, καταπίπτει. 103 εγκρίθηκε. Όχι, ωραία. Λοιπόν, 107 του κυρίου Επιτίδου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Α. Α, καταπίπτει. Εγκρίθηκε 9. Α, μάλιστα. Ωραία, 109 τότε. Υπέρ της 109 παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 του κυρίου Κόρβιν Μίκε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 103 δεν εγκρίθηκε. 111, 12 και 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 114. Καλώς.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 Πέρας. Απορρίφθηκε. 10 και 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 και 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ συγγνώμη την 126 μα η φιλελεύθερη είναι υπέρ. Μα είδα, είδα χέρια να σηκώνονται. Καλά, καλά. Ωραία. Να ελέγξουμε την 126. Πέρας. Απορρίφθηκε. Όλο εσάς κοιτάω. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 και 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Όχι. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές Η φιλελεύθερη είναι κατά, οπότε απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 και 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13, 140, 141, 142, 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές. Α, έτσι και αλλιώς καταπίπτει. 145 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 147 μέχρι 150 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται. Ας το επαληθεύσουμε. Ωραία, επαληθεύουμε. 147 ως 150. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτονται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14, 152, 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική πρόταση, wow, υπέρ, οι 7 κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά είχε. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Ωραία, επαληθεύουμε την 178. Αφού το έτοιμο έρχεται από το ΕΛΚ, να πω όχι. 198 Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις ακόμα απομένουν να ψηφίσουν. Λίγοι. Εγκρίνεται. Πού βρισκόμασταν. 179. Βαλέρο, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται.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 Η επόμενη καταπίπτει, πολύ ωραία. 192 υπέρ. Κατά εποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά εποχές. Επαληθεύουμε την 193. Λήξη. Απορρίπτεται. 194. Της κυρίας Βερζιά. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 196. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Κα, εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 197. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 199. κρυπαντζέρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. ...208. 204 έχει εγκριθεί, όχι. Συμβαστική 10. Α, υπέρ. Κατά. Εποχές. Η 10 εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 209 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 214 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21-22 υπέρ κατά εποχές. απορρίπτονται 23 υπέρ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 απορριπτώνται. 51 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. 51. Κύριο Παντζέρη. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη εγκρίνεται. Μαρίτια, με εκνευρίζει ότι μερικέ φορέ ψηφίζει ναι, αλλά έχει το δάχτυλό στον αντίχειρας προ τα κάτω. Ε, ίσως θα μπορούσα να σηκώσει μια σημαία, γιατί εγώ πραγματικά έχω πρεσβειοπία. Συμβαστική παρθυμόν 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. Αλλά οι φιλελεύθεροι ψήφισαν κατά σας. Σας βεβαιώνω. Τέλος πάντων. Επαληθεύουμε. Την 59. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. «62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Επαληθεύουμε. Την 63 έναρξη της ψηφοφορίας. Λείπουν ακόμα 5, 3... Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. με ναι, ενημερώνουν ότι θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την 65. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Και πάλι κυρία Βερζιά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Όχι, ναι, 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται η ο πρόεδρος. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την ομοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας ακόμη συνάδελφος κοιμάται. Λίγοι. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Λούνατσεκ. Έχουμε καθυστερήσει 20 λεπτά μετά από 100 λεπτά παραγωγικών ψηφοφοριών που απαιτεί ασφαλώς έξυπνους ανθρώπους. Περνάμε στο σημείο 17, ανταλλαγή απόψεων με τον Μεσιό Πατρικ Κι, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στην αεροπορία, της αεροπορίας. Καλωσορίσατε. Συγγνώμη που σας υποχρεώσαμε να περιμένετε μερικά λεπτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που, ο κύριος, ε, που υποδεχόμαστε τον κύριο Κι στην Επιτροπή μας. Πέρσι συμμετείχε σε μια ανταλλαγή απόψεων ε, στην ε, υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ και υπέβαλε έκθεση για την Ευρωπαϊκή Task Force για τις ζώνες σειράξεων που συνδεόταν με την πτήση 17 ε, των, της Malaysian Airlines. Η ασφάλεια σε πολλά μέρη του κόσμου και κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές των πολιτών μας όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η, ΙΑΣΑ υποστηρίζει την, ε, και την εξωτερική διάσταση της αεροπορίας μας, παίζει σημαντικό ρόλο Περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Κι, στον οποίο δίνω και το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που μιλώ ενώπιον σας σήμερα. Θα σας παρουσιάσω ποιοι είμαστε εν συντομία. Η αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες όταν ταξιδεύουν από αέρος και να τους προστατεύσουμε επίσης και περιβαλλοντικά. Γιατί η εντολή μας, η αποστολή μας μας υποχρεώνει να διασφαλίζουμε ότι οι κινητήρες και τα αεροπλάνα που παράγονται στην Ευρώπη είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης ε, πρέπει να εμπεδώσουμε την έννοια αγορά στην Ευρώπη μέσω κοινών κανόνων για την λειτουργία των αεροπορικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να προστατεύουμε τους ε, πολίτες μας σε όλο τον κόσμο. Και θα σας πω πώς το κάνουμε. Με μια ματιά ε, πριν από 15 χρόνια, είμαστε περίπου 800 άτομα με έδρα την κολονία και ε, γραφεία στις Βρυξέλλες. Έχουμε 32 μέλη, 28, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν 4 συνδεδεμένα μέλη, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενστάιν, 32 συνολικά. Ε, μία από τις ιδιαιτερότητες ε, της ΕΑΣΑ είναι ότι το 75, κατά 75% μας χρηματοδοτεί η βιομηχανία, ο κλάδος μάλλον. 30% περίπου από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό οι περισσότερες δραστηριότητές μας λαμβάνουν χώρα με τη στήριξη του κλάδου και σε συνεργασία με τον κλάδο. Ο διεθνή μας ε, ρόλος, και εδώ θα σας δώσω λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, ε, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω και στηρίζουμε τον κλάδο της ε, αεροπορίας στην Ευρώπη. Θα σας πω πώς το κάνουμε αυτό που κινούμαστε ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ασφάλεια της αεροπορίας προφανώς δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προωθούμε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Η αεροπορία είναι διεθνής δραστηριότητα εκ της φύσεώς της. Οπότε οπουδήποτε και να ταξιδεύουν οι πολίτες μας, οπουδήποτε και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Και βέβαια θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και δράση αν κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών μας. Δηλαδή, αν οι πολίτες μας ε, ταξιδεύουν με μια αεροπορική εταιρεία, οπουδήποτε και αν λειτουργεί, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, πληρεί τις προδιαγραφές. Και θα πρέπει να επιτηρούμε τις εταιρείε, τα αεροπλάνα τους κλπ. Και τέλος, θα πρέπει να στηρίζουμε τον κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως, συνάδελφοι. από την αντίστοιχη υπηρεσία των ΗΠΑ έχουν την εντολή να προάγουν ε, την, τον ηγετικό χαρακτήρα της, αεροπορικής, της αεροπορίας των ΗΠΑ στον κόσμο. Εμεί δεν έχουμε τέτοια εντολή, αλλά πρέπει να στηρίζουμε τον κλάδο σε όλο τον κόσμο. Σας δώσω με περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς στην πράξη επιτυγχάνουμε όλα αυτά. Πρώτον, πιστοποιούμε τα αεροπλάνα τα οποία χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές εταιρείες. Όχι μόνο η Airbus, αλλά και Boeing, Bombardier, μικρότερο σκάφη και στο μέλλον ενδεχομένως και ρωσικά και κινέζικα αεροσκάφη. Πιστοποιούμε όλους τις φορείς ε, που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες για την συντήρηση ε, όπως για, παράδειγμα ένα αεροπλάνο το οποίο ε, βρίσκεται σε μια χώρα στην Αφρική, εκεί συντηρείται από μια εταιρεία την οποία εμείς έχουμε πιστοποιήσει. Επίσης υποστηρίζουμε, ε, επίσης, ε, την, ε, τον κατάλογο ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφει τις μη ασφαλείς χώρες και αεροπορικές εταιρείες για τις οποίες εκδίδουμε συστάσεις στους Ευρωπαίους πολίτες να τις αποφεύγουν. Επίσης, εγκρίνουμε όλες τις τήσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από μη, ευρωπαϊκούς, ε, από μη ευρωπαϊκές ε, εταιρείες. Και τέλος, και έχουμε και έναν μηχανισμό έγκρισης σε ζώνες σειράξεων. Θα σας ενημερώσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Ήδη έχω ενημερώσει για την έκθεσή μας στην Επιτροπή. Ε, έχουν ε, στα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές επιθέσεις ε, εναντίον πολιτικών αεροσκαφών. Μετά λοιπόν από συζητήσεις με τα κράτη-μέλη συμφωνήσαμε έναν μηχανισμό που με την, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Home συλλέγονται όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα διάφορα κράτη-μέλη εντάσσονται στον Ευρω... ευρωπαϊκό μηχανισμό και ε, ανάλυσης και μετά εκδίδουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη για το κατά πόσο υπάρχουν ε, κίνδυνοι ή ε, απειλές. 16 τέτοιες ε, έχουν εκδοθεί τελευταία χρόνια Δεν είμαστε πολύ δημοφιλείς σε αυτές τις χώρες γιατί δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει πως δεν είναι ε, ασφαλείς χώρες. Παρ' όλα αυτά είναι καθήκον μας να το κάνουμε δεδομένου του ότι συνέβη στην Ουκρανία. Τι κάνουμε για την πρόθεση των ευρωπαϊκών προτύπων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε προγράμματα συνεργασία χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η ΕΣΑ τα διαχειρίζεται εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτών βοηθούμε διάφορα κράτη, κυρίω κυρίως το αναψώμενα κράτη, ε, να ε, ε, ανεβάσουν το επίπεδο ασφάλειας και προτύπων που χρησιμοποιούν. Πριν από 20 χρόνια είχαμε μόνο του κανονισμού των ΗΠΑ. Σήμερα βρισκόμαστε με τους δικούς μα κανονισμού βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ και ένα μεγάλο αριθμό χωρών έχει αποφασίσει να υιοθετήσει το 100% των, κανόνε αυτού και του κανονισμού. Ε, σας δείχνουμε ε, το χάρτη που βλέπετε ποιε είναι αυτέ οι χώρε. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε προφανώ έχουν υιοθετήσει αυτό το σετ κανόνων, αλλά βλέπετε ότι στην Νοτιοτελική Ασία, στην Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στην Κεντρική Αμερική έχουμε χώρε οι οποίε αποφάσισαν να υιοθετήσουν πλήρω τους κανόνες μας. Αυτό είναι καλό για το συνολικό επίπεδο ασφάλειας και σε αυτές τις χώρες αλλά και, στην, και για τον κλάδο μας. Και αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες ε, ε προορίζουμε ε, χρηματοδότηση για να τις βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στους κανόνες μας. Είναι μια πολύ επιτυχής προσπάθεια. Πολλές χώρες μας έχουν ζητήσει ε, βοήθεια για να αναπτύξουν περισσότερο και να εφαρμόσουν καλύτερα τους κανονισμούς μας. Στήριξη στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 80% των αεροπλάνων της Airbus πολλούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες IKEA, ICAO, ε, όλα τα αεροπλάνα τα οποία ε, εγγράφονται σε μια χώρα ταξινομούνται θα πρέπει να πιστοποιούνται σε αυτή τη χώρα και ε, για πολλές χώρες το θέμα αυτό είναι καθαρά γραφειοκρατικό, διοικητικό. Το να δέχονται τα πιστοποιητικά της ΕΑΣΑ, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία ε, έχει αποφασιστεί να πιστοποιούν τα προϊόντα μας προκειμένου ενδεχομένως να κερδίσουν και τεχνογνωσία για τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Εμείς στηρίζουμε τον κλάδο, στηρίζουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτέ πιστοποιήσει σε άσα. 130 ε, working arrangements, διευθετήσει εργασία, δηλαδή, υφίστανται με τρίτες χώρες που μας βοηθούν να συνεργαζόμαστε και να ε, πιστοποιούνται τα αεροπλάνα μας από αυτές τις χώρες. Υπάρχουν και τρεις αμοιβές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες για την αμοιβαία αναγνώριση με τον Καναδά, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται διμερείς συμφωνίες με την Κίνα και την Ιαπωνία. Επίσης συμμετέχουμε σε διεθνούς οργανισμούς τυποποίησης, διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Βλέπετε, βλέπετε εδώ, κάποιους από αυτούς. Πρέπει να πω ότι είμαστε λιγότερο ουδέτερο ισχυρή από τις ΗΠΑ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε άμεσα τι ε, διεθνεί αυτές οργανώσεις τυποποίηση. Οι ΗΠΑ την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης έχουμε ε, αντιπροσωπείες που στηρίζουν τον κλάδο. Βλέπετε σε ποιε πόλει Έχουμε τέσσερι αντιπροσωπείες με γραφεία στο Μόντρεαλ, την Ουάσιγκτον, στην Κίνα και τελευταία στη Σιγκαπούρη. Έχουμε πέντε άτομα, μόνιμο προσωπικό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, 120 έχει η Federal Aviation Administration των ΗΠΑ. Κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον κλάδο μας. τελευταίες μου κουβέντες το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εξυγχρονίζουμε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΑΖΑ. Υπάρχει ένας τριμερής διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπου περιλαμβάνεται διεθνής διάσταση, η οποία πρέπει να ενισχυθεί και βεβαίω μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά στα διεθνέ προσκήνιο. Σα ευχαριστώ για τη στήριξή σα, διότι είναι προς όφελος της ΕΑΖΑ και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μεσή. Ευχαριστούμε Κυριακή. Και τώρα να δώσω το λόγο σε συναδέλφους που θέλουν να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων. Πρώτος ο μιλητής, ο κύριος Δεγκράντες από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και ευχαριστώ τον κύριο Κι, τον επικεφαλής του ΕΑΣΑ. Αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι πάντα πολύ δημοφιλείς. Εμείς ως Κοινοβούλιο πάντα έχουμε κάποιες αμφιβολίες απριόρι και αυτό είναι αιτιολογημένο γιατί αυτοί οι οργανισμοί είναι μια προσπάθεια για να ε, χρηματοδοτηθούν εκτός προπολογισμού της Ένωσης ε, κάποιες δραστηριότητες. Αλλά εγώ έχω θετική ε, προσέγγιση. Και το έχω πει επανειλημμένα και στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου συμμετέχω εδώ και 12 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητος αυτός ο οργανισμός για να διασφαλίζεται η ασφάλεια στις ε, αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχει έκδεση Μαρινέσκου που συζητείται στον τριμερή διάλογο τώρα. Αυτός οπωσδήποτε θα μας ε, δώσει τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα αυτό, για το οποίο εργάζεται τόσο καλά. Εμείς έχουμε εκφραστεί επί του θέματος αυτού και όσο δεν αλλάξει θα συνεχίσουμε να εκφραζόμεθα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν δυσχέρειε για το άρθρο 2.6, για το Γιβραλτάρ το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινή λογική και για το 75 για την μεταφορά αρμοδιοτήτων η χώρα μου Ισπανία συμφωνεί μόνο αν έχει εθελούσια βάση αυτή η διάταξη και είμαστε και κατά των ε, τελών και είμαστε και κατά και των κατεξοδότηση πράξεων πρέπει κατά τη γνώμη μας μόνο να χρησιμοποιούνται για την ε, επικαιροποίηση του παραρτήματος για τα ντρόουν. Ευχαριστώ για όσα μας ε, παρουσιάσατε. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ο κύριος Μαρινέσκου θα ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω να ε, σας θέσω τα εξής θέματα. Πρώτον, ορισμένοι βουλευτές θέσαμε ένα ερώτημα και αναμένουμε απάντηση για τις μονομερές ενέργειες των Πολιτειών για τις ταμπλέτες και τα λάπτοπ στην ε, καμπίνα, στο αεροσκάφος δηλαδή, εντός του αεροσκάφους. Δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από τις συνηθισμένες χειρονομίες του Τραμπ ή αν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Αλλά εμείς διαφωνούμε. Γιατί αυτά είναι θέματα αρμοδιότητας της ΕΑΣΑ. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν συντονισμός, αν όχι εναρμόνιση. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται στην πολιτική αεροπορία τέτοιες αποφάσεις που μας στίγουν όλους και τους Ευρωπαίους, χωρίς να μπορέσουμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Ελπίζω να απαντήσετε. Άλλο θέμα. Μία άλλη έκθεση για την οποία είμαι και έχουμε θέσει το θέμα για την πιστοποίηση του εξοπλισμού για την ασφάλεια. Έχει μπλοκαριστεί το θέμα το Συμβούλιο. Το καταλαβαίνω βέβαια, γιατί σημαίνουν τεράστιο κόστος. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ότι στην παρούσα συγκυρία, όπου τα θέματα ασφαλείας είναι τόσο σημαντικά, είναι διατεθειμένοι οι πολίτες ακόμη να δεχτούν και περιορισμό των ελευθεριών τους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ε, μερική η προσέγγιση της Κομισιόν. Και ούτως ή άλλως αυτά που λέει η Κομισιόν θίγουν αρμοδιότητες του οργανισμού σας, του ΕΑΣΑ. Είμαι εισηγητής μιας έκθεσης πρωτοβουλίας για τις νέες τεχνολογίες. που μας δίνουν νέες τεχνικές δυνατότητες για να αυξήσουμε την ασφάλεια δεν υπάρχει πρόβλημα με τις τεχνολογίες. Υπάρχει πρόβλημα πόρων, υπάρχει πρόβλημα δέσμευσης για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ παραπλανητικό να πούμε, σε αυτή τη φάση, που είναι τόσο ευάλωτη η πολιτική αεροπορία σε αυτές τις απειλές, ε, υπάρχουν τόσο νέες μέθοδοι, τόσες νέες μέθοδοι τρομοκρατίας που προκαλούν ε, τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες από διάφορους τρομοκράτες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην κάνουμε τις αναγκαίες επενδύσεις για να υπάρχει η αναγκαία προληπτική ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Να εντάξουμε την ευρωπαϊκή μας αυτή πρωτοβουλία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Να το σημειώσει αυτό η Κομισιόν και να προωθήσει την πρότασή μας εντός διεθνών οργανισμών που μπορούν να προωθήσουν την παγκόσμια ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Αυτά τα θέματα ήθελα να θέσω, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν πολλές άλλες που σίγουρα θα θέσουν άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δεγκράντες. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Εάν απλώς σηκώσετε το χέρι σας, δεν έχουμε τόσο συχνά την ευκαιρία να έχουμε συνομιλία με τον κύριο Κι. Σπανίως συμβαίνει αυτό στην Επιτροπή μας. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο. Κύριε Κι, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Ντεγκράντες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξεκινήσω συζήτηση για τα σχόλια του Κοινοβουλίου εν του τριμερούς διαλόγου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποσυζήτηση έτσι κι αλλιώ. Για την απόφαση, την ενδεχόμενη απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν απαγόρευση για τις ε, προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές επί του αεροσκάφου, την καμπίνα του αεροσκάφου. Αυτή τη στιγμή το συζητάμε με την DFA τον ομόλογο φορέα της ΗΠΑ. Και μας απασχολεί το τι θα γίνει με τα λάπτοπ που μπορεί να μεταφέρονται στα αεροπλάνα. Οι μπαταρίες, όπως ξέρετε, έχουν την τάση διαρκώς να καίγονται από κάποιες συνθήκες. Θεωρούμε λοιπόν ότι όταν πρόκειται για ένα μεμονωμένο στοιχείο του λάπτοπ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν όλα τα λάπτοπ πάνε στην, ε, στις αποσκευές ε, του αεροσκάφους και φορτωθούν, θα κάνουν όλες οι μπαταρίες. Κοιτάζουμε λοιπόν τι μέτρα μπορεί να αναλυθούν, να ανακοινωθεί επισήμως η απαγόρευση Και το συζητάμε με τους ομολόγους μας από τις ΗΠΑ και άλλες γεωγραφικές περιοχές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό με φέρνει και στον αλληλοσυσχετισμό μεταξύ της ασφάλειας και της προστασίας. Όπως ξέρετε κύριε Δεγκράντες, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε σε όλα τα θέματα της προστασίας για να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Είναι πολλέ οι διεθνεί δραστηριότητε, όπω τα εργαλεία πιστοποίηση που αναφέρατε και το επίπεδο των απειλών δεν είναι το ίδιο για όλε τι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε. Άρα δεν μπορεί να είναι απλώ εθνική. Υπάρχει μάλλον και ένα μεγάλο κομμάτι εθνική αρμοδιότητα που έχει να κάνει με την προστασία. Όμω υπάρχουν κοινέ ευρωπαϊκέ απειλέ, κοινά ευρωπαϊκά έτε και κινητά. Συζητήσαμε για τις εμπόλεμε περιοχέ λόγω χάρη, όπου συμφωνήσαμε με διάφορες υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών ανά την Ευρώπη να ε, ενοποιήσουμε το πουλ πληροφοριών που διαθέτουμε και να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ασφαλή και την προστασία και τα σχετικά θέματα. Νομίζω ότι προχωρούμε σωστά. Η ανάλυση των απειλών και από την χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών στην καμπίνα του αεροσκάφου είναι ένα θέμα. Είναι σωστό λοιπόν η Ευρώπη να συγκεντρώνει τι πληροφορίε, να τι συλλέγει από κοινού για να μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κύ. Δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα σχόλια, άλλε ερωτήσει. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Και καλό ταξίδι πίσω στην κολονία. Ελπίζω να σα ξαναδούμε σύντομα. Ευχαριστώ. So, colleagues, we... Συνάδελφοι, μπορούμε τώρα να έρθουμε στο σημείο που αναβλήθηκε χθες το βράδυ. Απενημέρωση για την επίσκεψη στο Νότιο Κάφκασο, την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας. Όπως ξέρετε, έγινε μια ad επίσκεψη στο Σερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Αρμενία την περασμένη εβδομάδα, με συμμετοχή οκτώ μελών. Γήθηκα εγώ ίδιος ως πρόεδρος, οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου ήταν ο κ. Λάζλο Τέρκες, ο κ. Μαμίκιν από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, ο κ. Ζαμπάτσκι από του Συντατικού Μεταρρυθμιστέ, ο κ. Μπάιρ από του Φιλελεύθερου, ο κ. Σόλτζ από την ΚΟΕ και η κυρία Χάουταλα από του Πρασίνου. Η αντιπροσωπεία μα είχε ένα εντατικό πρόγραμμα, διότι ήμασταν μόνο τέσσερι μέρε εκεί για να επισκεφθούμε τρει χώρε και σε και στις τρεις χώρες συναντήσαμε τους πρόεδρους τους και υπουργού εξωτερικών και όλους τους αντιπρόεδρους των Εθνικών Κοινοβουλών. Ε, επίσης, τους πρόεδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων. Συναντήσαμε και ηγέτες κομμάτων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους πρεσβευτές των ευρωπαϊκών κρατών και ε, εργαζομένους σε διεθνείς οργανισμούς ασχοληθήκαμε με τα θέματα παρακολούθησης και εποπτείας και ε, στην Αρμενία αποτίσαμε φορό τιμή στα θύματα της γενοκτονίας στο ε, μνημείο του Γερεβάν και επισκεφτήκαμε και ε, μια σχολή ε, διαβίου κατάρτισης, επίσης, Είχαμε επίσης τέσσερις συνεντεύξεις τύπου και στην κάθε μια από τις τρεις αυτές χώρες. Η τελική μας δήλωση στον τύπο έχει δημοσιευθεί στο ιστοτοπό της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, χθες μόλις, και εντοπίζει τα βασικά ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή μα ε, στην επίσκεψή τη. Να τονίσω κυρίω για το Αζερβαϊτζάν. Η επίσκεψή μα ήταν απόδειξη ότι μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ε, Αζεριακού Κοινοβουλίου. Επίση, με τι διαπραγματεύσει για μια νέα συμφωνία συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλι ολοκληρωθούν αυτέ τι διαπραγματεύσει, θα μα ζητηθεί να δώσουμε και εμεί τη συγκατάθεσή μα. Ε, τονίσαμε ότι τα τμήματα τη συμφωνία πρέπει να βασίζονται σε κοινέ αξίε όπω η δημοκρατία, το κράτο δικαίου, η, η χρηστή κυβέρνηση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Και όλα αυτά είναι εξίσου σημαντικά όπω και το εμπόριο και οι τομιακές συνεργασίες. Ε, για την Γεωργία αποστήλαμε ένα σαφέ μήνυμα ότι είναι ε, πρωτοπόρο στην ε, γειτονία προ Ανατολά η Γεωργία. Τα βήματα πρώτα που έχουν γίνει είναι εντυπωσιακά και καλωσορίζουμε την πολύ θετική δουλειά για την υλοποίηση τη συμφωνία σύνδεση ταυτόχρονα. Ενθαρρύναμε την κυβέρνηση, την Διφλίδα, να συνεχίσει με τι προσπάθειε μεταρρύθμιση, ιδίω στον ε, τομέα των δικαστικών, την καταπολέμηση τη διαφθορά και την προστασία των μειονοτήτων. Τέλος, επαναεπιβεβαιώσαμε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ε, εθνική κυριαρχία της Γεωργίας και την εδαφική της ακυρεότητα. Και στην Αρμενία, το θέμα των Αγκόρνο Καραμπάχ ήθελε ε, ε, στην μέση κοιτάξη όλων των συναντήσεων και όπως και στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν, διαρκώς υπενθυμίζαμε την ευρωπαϊκή θέση επί του θέματος. Και παραθέτω εδώ, το status quo δεν μπορεί να διατηρηθεί, η ε, πόλεμη σύγκρουση δεν μπορεί να λυθεί στατιστικώ και χρειάζεται μια πολιτική λύση βάσει του διεθνού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει τι προσπάθειες διαιτησία και διαμεσολάβηση τη ομάδα ε, του ε, ΟΑΣΕ και Μίνσκ. Επίσης συζητήσαμε το θέμα με την Βουλή της Αρμενίας ε, ε, και την σχετική συμφωνία που προβλέπεται, ε, όπου θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει την συγκατάθεσή του. Είναι πάλι μια απόδειξη αυτό ότι η γειτονία προς Ανατολάς δεν είναι ένα παιχνίδι ανταγωνισμού με άλλους γεωγραφικούς πρωταγωνιστές εκεί. Συζητήσαμε και εκεί τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση των διακριτικών μεταχειρήσεων το επιχειρηματικό κλίμα πρέπει να δημιουργηθεί, καθώ και τα κίνητρα πρέπει να δοθούν για να τονωθεί η αποσχόληση ιδίω των νέων Αρμενίων. Είναι μια σοβαρότατη προσδοκία τη κοινωνία εκεί. Και με αυτά και με αυτά θα θέλω να δώσω τον λόγο στα μέλη τη αντιπροσωπεία μα εκεί και ε, ειλικρινώ και θερμό να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και του τρει πρεσβευτέ μα, την Πακού, την Τιφλίδα, την και το Κερεβέν. Ε, και τις ομάδες συνεργατών εκεί που προσέφεραν ε, εξαιρετική τεχνική στήριξη. Ε, ευχαριστώ επίση και για του πολιτικού συμβούλου μα τόπου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα τη γραμματεία τη ΑΦΕΠ για την εξαιρετική προετοιμασία και την πολύ καλή δουλειά που έκανε στι χώρε αυτέ. Αυτά από δική μου πλευρά θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου που συμμετείχαν στο ταξίδι μα. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Ζεύκο. Η κυρία Ζεύκο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι περιγράψατε με κάθε λεπτομέρεια την επίσκεψη που ήταν πολύ καταργανωμένη. Έχουμε τώρα μια πολύ καλύτερη εικόνα της κατάστασης σε αυτές τις χώρες και νομίζω ότι η επίσκεψη βοήθησε για να έχουμε πολύ στενότερες σχέσεις με τα κοινοβούλια και να περάσει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίξει περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Αντρέης Μαμίκινς. Εγώ θα μιλήσω τα λετωνικά που είναι πολύ γνωστά και στο Νότιο Κάφκασο. Οι Λετωνοί έχουν ε, παρουσία στην ε, Γεωργία από το 18ο αιώνα. δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά που είπατε. Η Γεωργία είναι η χώρα που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στο πρόγραμμα της Ανατολικής Γειτονίας. Ό,τι ζητήσαμε το έκανα. Όντως κάνουν ε, προσπάθειες. Ούτως ώστε η χώρα τους να προσεγγίσει όσο γίνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία, συμφωνώ με αυτά που είπατε Πρόεδρε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στο, στη σύραξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και θέσαμε το ερώτημα στον πρόεδρο της Αρμενίας και αυτό ε, μας έκανε να συζητήσουμε μαζί του για 40 λεπτά παραπάνω. Θέσαμε ένα ερώτημα που, από όπου βγάλαμε το συμπέρασμα ότι θα συνεχιστεί το αδιέξοδο για πολλά χρόνια ακόμη. Ξέρουμε ότι πρέπει να ισχύει η αρχή της εδαφικής ακαιρεότητας. Αλλά ο πρόεδρος της Αρμενίας είπε ότι κάθε χώρα πρέπει να επιλέγει τη μοίρα της και ότι μπορούν να δημιουργηθούν και καινούργιες χώρες. Οπότε είπα στον Πρόεδρο ότι στη Λετωνία το 1986 πολλοί μας λέγανε ότι δεν πρέπει να ονειρευόμαστε ανεξαρτησία, αλλά τελικά την αποκτήσαμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Θα συνεχιστεί το αδιέξοδο. πολύ διπλωματικοί έχουν τονίσει ότι είναι καλύτερα να έχεις 10 χρόνια διπλωματεύσεων από ε, μία μέρα πολέμου. Ευχαριστώ τώρα τον κύριο Σόλτς που επίσης συμμετείχε στην ε, αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ. Θέλω να ε, εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και προς τη γραμματεία μας και προς την αντιπροσωπεία μας επιτόπου που βοήθησαν πολύ το ιδιαίτερα περίπλοκο και πλήρες πρόγραμμα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Είναι σαφές ότι η διένεξη στον Αγκόνο Καραβάχ μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω ειρηνικών μεθόδων. Συζητώντας με διάφορους εκπροσώπους Συζητήσαμε και με εκπροσώπους των προσφύγων από το Αζερβαϊτζάν που είναι στην περιοχή του Μπακού. Είναι σαφέ ότι μόνο η ίδια η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί λύση. Δεν θα πρέπει να αρκεστούμε στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχών των χωρών αυτών ή και κάποιων ξένων διπλωματών. Πρέπει να αυξηθεί συνειδητότητα, συνειδητοποίηση μάλλον, του ότι οι ίδιες οι κοινωνίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ιδιαίτερα μακροχρόνιο πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι ε, ε, παρόμοια και στην ε, Οσετία και την, την Νότια Οσετία και την Απχαζία. Συναντηθήκαμε παντού και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση των πολιτικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και του δικαστικού συστήματος αλλά εγώ ε, και ίσως και άλλα μέλη της αντιπροσωπής να συμφωνούν σε αυτό που θα πω ότι ορισμένες φορές είχαμε την εντύπωση ότι δεν είναι ιδιαίτερα ριζωμένοι στην ε, κοινωνία τους. Σε τι βαθμό αυτοί οι εκπρόσωποι των οργανώσεων συνδέουν συνδέουν την καθημερινή τους εργασία με την καθημερινότητα των ε, ανθρώπων, των πολιτών των χωρών. Βεβαίως προσπαθούν να προωθήσουν ε, τα διεθνή πρότυπα, τις αξίες της δικές μας για κοινωνικά θέματα, για περιβαλλοντικά θέματα. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Η Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τον ε, εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο ηγηθήκατε αυτής της αντιπροσωπής και ήταν πραγματικά προνόμιο η συμμετοχή μου σε αυτήν την αποστολή. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για όλους μας για να αποκτήσουμε μια ιδέα για την ε, κατάσταση και των τριών χωρών. Βεβαίω η καθεμία έχει τα προβλήματά της. Εγώ θεωρώ ότι το Αζερβαϊτζάν που τώρα ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις για την ειδική εταιρική σχέση θα πρέπει να κατανοήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τονίσει την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η επίσκεψή μας συνέπεσε με την ε, τρίτη επέτειο από, με, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Μαμάντοφ που είναι ακόμη στη φυλακή παρά το ότι το δικαστήριο αυτό αποφάσισε ότι θα έπρεπε να απελευθερωθεί και δεν είναι ο μόνος πολιτικός κρατούμενος. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέσει προϋποθέσεις για την διαπραγμάτευση αυτής της νέας σχέσης. Για την Αρμενία η νέα συνολική ενισχυμένη εταιρική σχέση ήδη λειτουργεί και μέσω της εφαρμογής ελπίζω να ενθαρρύνουμε την Αρμενία να προωθήσει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατία τώρα που περνάνε σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα που οπωσδήποτε προωθεί την, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ήμουν ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας παρατήρησης των τελευταίων εκλογών και ελπίζω η ΕΕΣ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να τονίζουν ότι ναι με ένωση ένωση επενδύσαμε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στην, ε, στον εξοπλισμό για τις εκλογές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτά που συμβαίνουν εκτός των εκλογικών τμήματων. Πρέπει να υπάρξει μια ορίμανση της ε, πολιτικής κουλτούρας. Δεν πρέπει να υπάρχει αγορά ψήφων και προσπάθειες εκφοβισμού. Τώρα για τη Γεωργία βεβαίως είναι η χώρα που ηγείται των προσπάθειών μας. Ε, πρέπει όμως να προσέχουμε γιατί πριν από λίγο καιρό η Μολδόβα ήταν ε, η ηγετική χώρα και βλέπουμε τι έγινε εκεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν οι αναγκαίες δικαστικές μεταρρυθμίσεις στη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χαϊντή. Για την άλλη, ο κύριος Χαγερνάτη. Η σύγκρουση στον Κάφκασο έχει συνέπειες που ξεπερνούν την, τα σύνορα της περιοχής αυτής ο πόλεμος των Αγκόρνο Καραμπάχ ε, θα πρέπει να ειδωθεί ε, ως προς τις αιτίες της. Ε, τον Αγκόρνο Καραμπάχ τεχνικά και πολιτικά ανήκει στο Αζερβαϊτζάν. Ε, συνεπώς με βάση την αρχή της ε, ε, ε ενότητας ε, όπως και η Οσετία στη Γεωργία ανήκει στο Αζερβαϊτζάν όμως όταν το κοσυφοπέδιο ε, διέριξε τη συνθήκη του Ελσίνκη η Ρωσία και κάποιες άλλες από τις ευρωπαϊκές χώρες είχαμε πει ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας ε, όταν ε, ανεξαρτοποιήθηκε η Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν η, το, του Ναγκόρνο Καραμπάχ συγγνώμη και της Οσετίας διορθώνει ο μιλτής, ε, είπαν ότι αυτές οι, δύο, οι δύο αυτές περιοχές είπαν ότι δεν ήθελαν να δεχτούν να αποτελέσουν τμήμα του Αζερβαϊτζάν και της Γεωργίας. Στην διαδικασία του Μίνσκ, όπου η Γαλλία, οι και η Ρωσία είναι οι τρεις βασικές ε, ε, χώρες σε ό,τι αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, ε, υποστηρίζουν ότι μέσω μιας διαδικασίας ανακοχής, απόσυρσης των στρατευμάτων ε, κλπ. Ε, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το καθεστώ του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα πρέπει να το αποφασίσουν οι δικατικοί του. Δηλαδή για δεύτερη φορά καταργείται το Ελσίνκι και δημιουργείται η αρχή της αυτοδιάθεσης ε, που υπερβαίνει την αρχή της, ε, ε, της εδαφικής Αναρωτιέται λοιπόν κανείς ε, πόσα σταθμά χρησιμοποιούμε. Αν τα αυτόνομα κοινοβούλια της Οσετίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ ε, έθεσαν το προηγούμενο ε, της απόσχησης γιατί ε, δεν δεχόμαστε για την Οσετία αυτό που δεχόμαστε για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και αν εφαρμοστεί για την Οσετία, γιατί όχι και στην Κρυμαία. Η διαδικασία αυτή είναι ε, κατ' εξαίρεση επαναστατική και γενικεύει μία συγκεκριμένη ε, περίπτωση που εφαρμόστηκε για μία πολύ μικρή περιοχή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις περιπτώσεις. Ε, η Ρωσία λέει τι χρειάζεται η Δύση 2.000 ε, νεκρού στην Κρυμαία για να δεχτεί αυτό που δέχεται στον Αγκόνο Καραμπάχ πως είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση συνένεση στον Αγκόνο Καραμπάχ που μας οδηγεί σε ακρότητα στην Κρυμαία τα θέματα αυτά είναι παγκόσμια δεν μπορούν ε, να ειδωθούν ε, κατακαιρματισμένα το Αγκόρνο Καραμπάχ λοιπόν, είναι, στον Αγκόρνο Καραμπάχ σημαίνει αυτό που θα συμβεί και στην Κρυμαία. Και πάλι θα καταγγείλουμε ε, ε την προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά το έχουμε ξεκινήσει από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ευχαριστούμε κύριε Νάρτ για τη συνεισφορά σας εσάς και όλους τους υπολείπους. Ως να την μέρος για την αποστολή μας, άλλα σχόλια. Κύριε Γκάλε, πολύ γρήγορα. Ναι, στην Γεωργία είχατε την εντύπωση ότι οι όλες οι συζητήσεις για την συνταγματική ε, μεταρρύθμιση δείχνουν να υπάρχει κάποια ε, πλειοψηφία που να αναδύεται, που να ξεπερνά τα δύο τρίτα του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης. Βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια βάρκα ή υπάρχει αντιπαράθεση για την συνταγματική μεταρρύθμιση. Το θέμα της συνταγματικής μεταρρύθμισης συζητήθηκε όχι μόνο με εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά κυρίως με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επίσης, συναντήσαμε τρεις ομάδες της αντιπολίτευσης, τρία κόμματα. Το Ευρωπαϊκό Όνειρο, την Ενωμένη Γεωργία και το άλλο ποιο τα πατριώτες για τη Γεωργία, υπέρ της Γεωργίας. Ναι, είδαμε να υπάρχει ευρία συνένεση. Και όχι μόνο προ τη συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά και του εκλογικού συστήματος του εκλογικού νόμου. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θέλουν να εργαστούν ε, ε, μαζί για τις βασικές αρχές. Κάτι που θέλετε να προσθέσετε για τον εκλογικό νόμο, βεβαίως, συστήσαμε ε, θερμό στις ε, στις αρχές της Γεωργίας να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Νομίζω κάποιοι επιφυλάσσονται περισσότερο από άλλους και διστάζουν περισσότερο από άλλους να το κάνουν αυτό. Έτσι. Χάιντι. Ε, ναι, μια κουβέντα. Εγώ βρήκα ότι είναι πολύ αποσχολημένο ότι το νέο κοινοβουλίο ήδη πριν τα Χριστούγεννα είπε ότι ε, είναι ταγμένο στην ε, ε, τήρηση των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας. Δεν ξέρω αν αυτό καλύπτει όλε τι του πολιτικού βίου, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική υπόσχεση. Ευχαριστώ. Και άλλη μια κουβέντα. Βεβαίως, το ταξίδι των τριών συναδέλφων στον Αγκόνο Καραμπάχ ήταν θέμα και στι συνεντεύξει τύπου, όχι μόνο στην Πακού και στο Κερεβάν. Και στι δύο συνεντεύξει τύπου είπα ακριβώ τα ίδια πράγματα, έδωσα την ίδια απάντηση. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου είναι ελεύθερα να ταξιδεύουν, μπορούν να κάνουν λίγο πολύ ό,τι του αρέσει, Όμω αυτοί οι τρει συνάδελφοι που πήγαν στον Αγόρνο Καραμπάχ δεν είχαν δικαίωμα ούτε καν να δηλώσουν κάτι, να εκφραστούν εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πήγαν ω ιδιώτε και υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να υποστούν τι συνέπειε που ενδεχομένω να έχουν. Γνωρίζετε ότι όχι μόνο εγώ αλλά και η κυρία Χάουταλα και ο κύριο Καρύμ απευθύναμε επιστολή προ το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και τη Αρμενία για την επισκέψη μα εκεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην συνεδρία στο Διευρυμένου Προεδρείο. Πριν το κάνω αυτό, να σας πω απλώς για το σημείο 20, η επόμενη είναι στις 19 Ιουνίου από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα και στις 20 Ιουνίου από τις 9 στις 10.30 και 3 και 6.30 στις Βρυξέλλες.